Καλημέρα Elnök. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι! ξημερώνει μια καινούργια μέρα, η τελευταία μέρα της τελευταίας Συνόδου Ολομελίας στο Στρασβούργο για το 2016. Θα συζητήσουμε την πρώτη έκθεση της ημερήσιας διάταξης που αφορά